il presidente buongiorno Γεια σας, αρχίζουμε τις εργασίες μας. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι τα πρακτικά από εχθές ε, έχουν ήδη διανεμηθεί. Αν δεν έχετε παρατηρήσει από αυτόν, τα πρακτικά εγκρίνονται πήραμε από τις ε, πολιτικές ομάδες, από τους σοσιαλδημοκράτες και από τους χριστιανδημοκράτες κάποιες, ε, κάποια αιτήματα για αλλαγή ε, των επιτροπών και τα ονόματα θα εμφανιστούν αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τα πρακτικά. Αυτές οι προτάσεις θεωρούνται δεκτές εγκεκριμένες. Πάμε τώρα στην ε, παρουσίαση του Συμβουλίου για να μας ενημερώσει για τη Ρουμανική Προεδρία. Και θα ήθελα να ενημερώσω τους ευρωβουλευτές ότι ε, αυτή η διαδικασία, αυτή η συζήτηση δεν είχε ε, προβλεφτεί, δεν θα ακολουθήσει κατζιάι, ούτε θα γίνουν δεκτές μπλε κάρτες. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Πρωθυπουργό, την κυρία Τάντσιλα, η οποία είναι κοντά μας στην Ολομέλεια να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από τη Ρουμανική κυβέρνηση να δώσω το λόγο στην κυρία Πρωθυπουργό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ενώπιον ε, του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω τον απολογισμό της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναν απολογισμό που περιέχει και σημεία αναφοράς για τον κοινό ευρωπαϊκό δρόμο που είναι μπροστά μας. Ως πρώην μέλος αυτού του σώματος γνωρίζω και ε, εκτιμώ τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς ήδη ε, έχετε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ με πολλή επιτυχία και στην ε, ε, εκτέλεση της θητείας σας. Κυρίε και κύριοι, ήταν σημαντικό να δείξουμε ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν για τους πολίτες και ιδιαίτερα ότι έχουν αποτελέσματα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και προσφέρουν προοπτικές για το μέλλον. Ε, με ικανοποίηση δηλώνω ότι η Ρουμανία πέτυχε αυτό το πράγμα. Αναλάβαμε αυτή την ευθύνη ως αποστολή προς τους πολίτες και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρήσαμε απαραίτητο, πως όλες οι δράσεις μας, να οικοδομούνται γύρω από την συνοχή ως κοινή ευρωπαϊκή αξία. Η Ρουμανία κατέδειξε ότι μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία ε, και να αντιμετωπίσει προκλήσεις και τάσεις ε, που θέτουν σε αμφισβήτηση την, ε, τον δρόμο της Ευρώπης. Αποδείξαμε ότι η δυνατότητα της Ρουμανίας να συμβάλλει στην προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που φαίνεται στον απολογισμό τον οποίο παραδίδουμε. 90 νομοθετικά εισφακέλους που κλείσαμε και σχεδόν 2.500 εκδηλώσεις, συναντήσεις και συνέδρια που οργανώθηκαν. Ταυτόχρονα διευκολύναμε την έγκριση 84 ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίων σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος επιθυμήσαμε με την εκτέλεση αυτή της εισιτηρία να έχουμε ορατά αποτελέσματα, η φορά βιώσιμα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να αναφέρονται εύκολα σε αυτά και με σαφήνεια. Αυτά τα αποτελέσματα ε, δίνουν μια αξιόλογη ε, ταυτότητα της πρώτης δικής μας προεδρίας που θεωρώ ότι μπορούμε όλοι να αναφερθούμε. Για παράδειγμα, θα ήθελα να πιστεύω ότι όταν ένας, Ρουμάνος, ε, ένας Ευρωπαίος πολίτης θα έχει καλή ισότιμη πρόσβαση και πιο ε, διαφανή πρόσβαση στο χώρο εργασίας που να του δίνει τη δυνατότητα να ισορροπεί την επαγγελματική ζωή με την ιδιωτική ζωή, θα ξέρω ότι αυτές οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Επίσης, θα ήθελα να πιστεύω ότι ο Ευρωπαίος πολίτης θα νιώθει σε μεγαλύτερη ασφάλεια, πιο προστατευμένος εντός των συνόρων της Ένωσης χάρη στις προσπάθειες της δικής μας Προεδρίας. Κατορθώσαμε να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα προς αυτή την κατεύθυνση. Από εδώ και μπρο θα είναι δυνατόν να γίνουν πιο αποτελεσματικές επαληθεύσεις στα εξωτερικά σύνορα, θα βελτιώσουμε την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας. Εξασφαλίσαμε σταθερά αποτελέσματα και στους τέσσερις πυλώνες προτεραιότητες της Προεδρίας.